τρίτες χώρες. Η τεχνολογία μας να μην εξαρτάται από τρίτες χώρες. Η συνεργασία θα βοηθήσει σε αυτό. Η μείωση της τεχνολογικής μας εξάρτησης είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φακέλου αυτού. Και είμαι σίγουρη ότι η άμυνα θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μιλάμε ακόμα για την ε, αμυντική βιομηχανική συνεργασία. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται για την συμφωνία ε, στην οποία καταλήξαμε μετά τους τριμερείς διαλόγους. Και ελπίζω αύριο να υπερψηφιστεί η πρόταση αυτή. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ όλους, τον εισηγητή, τους και όδες εισηγητές, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε, τον κύριο Μπούτσεκ, γιατί είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σκληρή δουλειά. Δεν ήταν εύκολο, αλλά νομίζω ότι η συμφωνία είναι ικανοποιητική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο ε, και τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης η οποία κατέδειξε ότι δεν συμβίπτουν οι απόψεις μας. Στους σοσιαλδημοκράτες ε, εκφράστηκαν από πλευράς τους διαφορετικές απόψεις ε, και στο επίπεδο των, στο μέτωπο των πρασίνων και εκεί διαφορετικές απόψεις. Ε, υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Υπάρχουν κράτη όπου δεν υπήρξαν εισβολές ε, ούτε κατοχή εδαφών. Από την άλλη όμως υπάρχουν κράτη όπως οι χώρες της ε, Βαλτικής ε, και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που εξακολουθούν να αισθάνονται υπό απειλή. Ναι, καλά τα κοινωνικά προγράμματα, αλλά αν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία, τότε προφανώς και κινδυνεύει η κοινωνική μας ευημερία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Αυστριακή και τη Ρουμανική Προεδρία γιατί δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και ε, επέδειξαν ε, ιδιαίτερη τεχνογνωσία και όσοι φοβούνται το θέμα των σχέσεων με τον ΝΑΤΟ, να τους πω το εξής. Κοιτάξτε, στη δική μας την περιοχή ξέρουμε πολύ καλά τι είπατε. Είμαστε υπέρ αυτού του ταμείου, αλλά είμαστε και υπέρ του ότι το ΝΑΤΟ εγγυάται την ασφάλειά μας. Είναι ο εγγυητής της ασφάλειάς μας. Επ' αυτού δεν αλλάζει τίποτα. Και θα θέλαμε άλλες χώρες, η Γαλλία παραδείγματος χάρη, να δραστηριοποιηθεί για την προστασία της ε, ανατολικής πτέρυγας ε, του ΝΑΤΟ. Ε, τέθηνε ερώτημα ε, από τι ή πώς θα ωφεληθεί η Πολωνία. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορούμε αν συνεργαστούμε να εξυγχρονίσουμε τον, ε, τους εξοπλισμούς, τη βιομηχανία εξοπλισμών ε, και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω ε, τα κονδύλια αυτού του ταμείου να διατεθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι άλλο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υπερψηφίσετε το κείμενο ε, όπως ακριβώς ε, το διαπραγματευτήκαμε. Παρακαλώ να απορρίψετε όλες τις τροπολογίες υπέρ του 31CP και υπέρ όλων των ε, τροπολογιών της Ολομέλειας, γιατί αλλιώς θα καταπέσει η συμφωνία μας. Αυτή είναι η θερμή μου παράκληση προς όλους σας. Το γεγονός αυτό, όπως σας είπα, το έχω ενστερνιστεί, γιατί αποτελεί ευκαιρία για την αμυντική βιομηχανία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και για την βελτίωση των αμυντικών μας ικανοτήτων που είναι πολύ σημαντικές. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να επερασπιστούμε τον τρόπο ζωής μας και τον πολιτισμό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, συγχαίρω και ευχαριστώ τον ομιλητή. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Τώρα προχωράμε. Κοινή συζήτηση για τα καλυμμένα ομόλογα. Έκθεση του κυρίου Μπέρντ Λούκε και θα ακολουθήσει και μία άλλη συζήτηση για τα καλυμμένα ομόλογα και τα, η δημόσια εποπτεία. Είναι δύο εκθέσει του κύριου Λούκε. Κύριε Λούκε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για κάθε αγορά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ασφαλή, ασφαλείς κινητές αξίες. Γνωρίζουμε δυστυχώς βέβαια ότι αυτό σπανίζει. Γνωρίζουμε ότι οι τιτλοποιήσεις δεν προσφέρουν επαρκή κάλυψη. Αυτό το γνωρίζουμε το αργότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι και τα κρατικά ομόλογα δεν προσφέρουν επαρκή προστασία. Ούτε και αυτά της Ευρωζώνης δεν είναι ικανοποιητικά ασφαλή. Όπως σας είπα, το συνειδητοποίησαμε και με την κρίση του ευρώ και του δημόσιου χρέους. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν ε, τα καλυμμένα ομόλογα, ότι αυτά είναι ασφαλή τα καλυμμένα ομόλογα υπάρχουν εδώ και πάνω από 250 χρόνια και μέχρι τώρα ε, δεν έχουν καταρρέψει. Πρόκειται για μια κινητή αξία που την χρειαζόμαστε στην Ευρωζώνη και στην κεφαλαγορά. Γι' αυτό λοιπόν εκπλήσει το γεγονός ότι τα καλυμμένα ομόλογα δεν έχουν εξελιχθεί επαρκώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι υπάρχει μόνο μία μικρή ομάδα κρατών που έχουν αυτή την παράδοση των καλυμμένων ομολόγων και την χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν σχεδόν καθόλου εμπειρία από καλυμμένα ομόλογα και δεν έχουν και σχεδόν καθόλου νομοθεσία για αυτά. Αυτό προσπαθούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε εκδίδοντας ή ε, θεσπίζοντας, ψηφίζοντας οδηγία και κανονισμό για τα καλυμμένα ομόλογα. Η οδηγία είναι παράλληλα και το οδηγό νήμα για τις εξελισσόμενες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με τα καλυμμένα ομόλογα επιτυγχάνουν και αποκτούν ένα αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, μπορούν να μεταφέρουν στην νομοθεσία τους αυτό που έχει αποδειχθεί σωστό εδώ και πολύ καιρό και που είναι μια πρακτική, δοκιμασμένη πρακτική στο θέμα των καλυμμένων ομολόγων. Όσον αφορά τη νομοθεσία, πραγματικά προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όλα αυτά που αναφέρουμε, που πιστεύουμε για τις κινητές αξίες, όλα αυτά ε, για τα οποία διαπραγματευτήκαμε και νομίζω ότι τελικά καταλήξαμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η οδηγία για τα καλυμμένα ομόλογα έχει τώρα λάβει τέτοια μορφή έτσι ώστε να έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες καλυμμένων ομολόγων. Αφενός εκείνα τα καλυμμένα ομόλογα τα οποία ορίζονται στον κανονισμό ε, περί επάρκειας κεφαλαίων, ομόλογα τα οποία προσέλκυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι είναι τα καλυμμένα ομόλογα υπό εξέλιξη, εκείνα που θα προσφέρουν νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, θα εξετάσουν νέες δυνατότητες εξασφαλίσεων. Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ καλές συνθήκες πλαίσιο, έτσι ώστε τα καλυμμένα ομόλογα να επικρατήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ικανοποιητικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο και αυτές οι κινητές αξίες να γίνονται αποδεκτές και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε να θέσουμε πρότυπα σε διεθνές επίπεδο για αυτό το χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Θα μπορέσουμε να τραβήξουμε την εμπιστοσύνη των ε, ε, πιστωτών και των ομολογιούχων. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και το ενδιαφέρον των οντοτήτων, ε, των εκδότριων οντοτήτων, έτσι ώστε να να ανοίξει η αγορά μας και να μην κλείσει έναντι εκείνων οι οποίοι επίσης ενδεχομένως ενδιαφέρονται για τη χρήση αυτού του εργαλείου. Νομίζω ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σήμερα. Προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία και βεβαίω θέλω να ελπίζω ότι αυτό το εργαλείο θα γίνει ευρέω αποδεκτό στην Κεφαλαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τώρα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Μπιερκόφσκα, παρακαλώ. μικρόφωνα, παρακαλούμε. Τα καλυμμένα ομόλογα είναι μια σταθερή πηγή και αποτελεσματικέ προ το κόστο πηγή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια τη κρίση. Ανταποκριθήκαν καλά. Είναι πάρα πολύ δημοφιλή σε κάποια κράτη-μέλη, ενώ σε κάποια είναι κάτι καινούριο. Η πρόταση τη Κομισιόν προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω αυτή την αγορά, βασιζόμενη στα υψηλά πρότυπα και τι καλέ πρακτικέ των εθνικών συστημάτων. Πρόκειται για ένα βασικό ε, στοιχείο τη. Ε, αγοράς Κεφαλογορών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πανευρωπαϊκή αγορά ομολόγων που θα υποστηρίζει το δανεισμό στην πραγματική οικονομία χωρίς να ενοχλεί ήδη τις εθνικές αγορές που λειτουργούν καλά. Θα υπάρξει όθηση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων στα κράτη-μέλη όπου είναι λιγότερο αναπτυγμένες αυτές οι αγορές. Οι κανόνες αυτές ε, θα σημαίνει ότι ε, θα υπάρχουν ασφαλή εργαλεία για τις τράπεζες που θα επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουν τις εταιρείε και τα Κυριά. Εκτιμούμε ότι η πεθανή εξοικονόμηση για τους δανειστές θα είναι περίπου 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης, θέλει η Ένωση να εναρμονίσει τους κανόνες προληπτικής εποπτείας προκειμένου να συνεισφέρουμε στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε δύο πυλώνε. Καταρχήν σε μια οδηγία που παρέχει ένα κοινό ορισμό των καλυμμένων ομολόγων, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των μέσων και εντοπίζει ε, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλή ποιότητα που μπορούν να επιλεχθούν για να καλυφθούν από καλυμμένα ομόλογα. Επίση, έχουμε και την οδηγία για την εποπτεία ε, και θέτει του κανόνε για τι ε, ετικέτε. Και ο δεύτερο νομοθέτημα, ο κανονισμό ενισχύει του κανόνε για πρώτα μισή εργασιακή μεταχείριση που θα, που θα καλύπτουν τα ομόλογα που αγοράζονται από τράπεζε. Όπως ε, είδαμε στους τριμμένους διαλόγους και έχουμε και στη δήλωση της ε, Κομισιόν, η Κομισιόν θέλει να τροποποιήσει την ε, αναλογία για την κάλυψη ρευστότητα για να ρυθμίσει τα καλυμμένα ομόλογα. Αυτό θα, καλύψει, θα αντιμετωπίσει συγγνώμη, την επικάλυψη μεταξύ του ε, του αποθέματος ρευστότητας ε, αποθέματος αλλιές για τα συνολικά στοιχεία. Ε, θα στείλουμε αυτά τα στοιχεία στο Κοινοβούλιο πριν από την ευρενή ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την επιτυχή για το επιτυχές αποτέλεσμα και κυρίως τον εισηγητή και όλους τους κοιόδες εισηγητές. Ο στόχος της πρότασης της Κομισιόν διατηρούεται χάρη στην επικοδομητική προσέγγιση της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου και της καλής συνεργασίας με το Συμβούλιο. Η μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο και εφαρμογή των νέων κανόνων για τα καλυμμένα ονόλογα θα πρέπει τώρα να προχωρήσει γρήγορα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι έχουμε μια σημαντική πηγή χρηματοδότηση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη προωθώντα τις ε, θέσεις εργασία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ροζάτη. Παρακαλώ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εργαζόμαστε πάνω σε δύο έγγραφα, τα οποία δημιουργούν νέες αρχές λειτουργίας για τα καλυμμένα ομόλογα. Πρόκειται για εγγυημένα ομόλογα και είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο δημιουργεί μια κεφαλιακή ένωση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό. Αυτά τα εγγυημένα ομόλογα ορίζονται το ορισμό του στο έγγραφο αυτό. Και τι είναι, είναι μια εγγύηση. Επίσης έχουμε δύο κατηγορίες εγγύσεων. Έχουμε τις ευρωπαϊκές που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και έχουμε τις premium, οι οποίες επιπλέον καλύπτουν και τις απαιτήσει του κανονισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, του CRR. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί από μόνη της να αποφασίσει για το πούλο του ενεργητικού και για το ρευστό. Καταλήξαμε σε ένα συμβασμό το 8% εγγύσεων για την ποιότητα των πιστώσεων. Επίσης υπάρχουν οι τραπεζικές εγγύσεις που γίνεται ένα εγγραφό υψηλής ποιότητας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον ε, βουλευτή, τον Ευρωβουλευτή Λούκε για την εξαιρετική αυτή έκθεση, αλλά επίσης και για την καλή συνεργασία που είχαμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική της συμμετοχή. Ζητώ από όλους τους ευρωβουλευτές να υπερψηφίσουν χωρίς τροπολογίες αυτή την έκθεση. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Σαντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς για τα καλυμμένα ομόλογα, όπως ονομάζονται. Η διαδικασία ξεκίνησε εδώ το 2017 με μια έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία θέσε και τις βάσεις του έργου μας για το νομοθετικό πακέτο που σήμερα έχουμε μπροστά μας. Δεν ήταν εύκολο, γιατί στην κάθε χώρα τα καλυμμένα ομόλογα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Αποτελούν ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του κατά τους αιώνες έχουν βέβαια αναπτυχθεί διαφορετικά στις διάφορες εθνικές αγορές, αλλά έχουν νόημα. Και σε κάποιες αγορές όπως τη Δανία και τη Γερμανία τα καλυμμένα ομόλογα θεωρούνται ένα μέσο επενδυτικό πάρα πολύ συνηθισμένο. Σε άλλες χώρες όπως τη δικιά μου τη Μάλτα δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχει εδώ λοιπόν μια πολιτική πρόκληση μπροστά μας για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην ε, αγορά, ε, την, ε, μάλλον την ένωση της κεφαλαϊκής αγοράς. Ε, θα έπρεπε όμως να αποφασίζονται όλα από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ή θα έπρεπε να δεχτούμε τις διευθετήσεις που έχουν γίνει στις εθνικές αγορές μέχρι τώρα και που έχουν αποδείξει την αξία τους. Εγώ θα συμφωνούσα με το δεύτερο. Ε, δεν πρέπει να αλλάξουμε πράγματα τα οποία έχουν λειτουργήσει για δεκαετίες, για αιώνες ε, ικανοποιητικά. Βέβαια, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να δημιουργηθεί με στόχο την προδευτική σύγκληση προς παρόμοιους κανόνες και πρακτικές. Το σεβαστικό κείμενο που έχουμε μπροστά μας ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή την πρόκληση. Περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής ΕΚΟΝ του 2018 και διορθώνει διάφορες πτυχές που θα ήταν μια ανησυχία για την ομάδα μου. Το κείμενο λοιπόν προωθεί την αναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενισχύει την διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών, ενώ συγχρόνω αποφεύγει τον κίνδυνο ανατροπή των επιτυχημένων εθνικών συστημάτων καλυμμένων ομολόγων. Χαίρομαι που αυτέ οι προτεραιότητε αντικατοπτρίζονται στο κείμενο και κάνω έκκληση στο Σώμα να εγκρίνει αυτήν την πρόταση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ, ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Πόση ώρα έχω κύριε Πρόεδρε. How much time I have, Mr. Chairman? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. 30 seconds. Thank Και 30 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη υπάρχει έντονος σκεπτικισμός για αυτού του είδους τα ομόλογα όταν φυσικά έχουν δει όλοι ότι ακόμη και κρατικά ομόλογα έχουν καταρρεύσει. Ιδίως στην πατρίδα μου όπου τα ελληνικά κρατικά ομόλογα τα οποία εμπιστεύτηκαν οι έλληνες πολίτες πάρα πολλοί μικρομεσαίοι συνταξιούχοι επένδυσαν τις, ε, τους κόπους μιας ζωής στα ελληνικά ομόλογα και ήρθε μετά το περίφημο psi με απόφαση του eurogroup και κουρεύτηκαν τα ομόλογα αυτά κατά 53%. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι στην Ελλάδα που είχαν εμπιστευτεί τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που δεν έχουν πλέον χρήματα να πληρώσουν τα φάρμακα να μπορέσουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο. αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουν καταρρεύσει τα κρατικά ομόλογα υπάρχει δυσπιστία απέναντι σε αυτή τη μορφή ομολόγου και φυσικά όπως αναφέρει στην εισήγησή του ο κύριος λούκε κάνει προσπάθεια η εισήγηση αλλά βεβαίως και ο κανονισμός να υπάρξουν οι μέγιστες εγγυήσεις ούτως ώστε αυτά τα ομόλογα να θεωρηθούν ασφαλή να έχουν φυσικά και πολλούς επενδυτές και έτσι να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο το οποίο θα διαμορφώσει μια συνολική αγορά και ταυτόχρονα θα πάρει κοντά του και αρκετούς επενδυτές. όμως θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα γίνουν αυτές οι διασφαλίσεις ούτως ώστε πραγματικά να μην φτάσουμε σε σημείο να καταρρεύσουν ακόμα και αυτά τα ομόλογα. όλα φυσικά κρίνονται από το πώς θα λειτουργήσει η αγορά. αν υπάρχει μεγάλη κρίση τότε πολλοί διερωτώνται αν και αυτά τα ομόλογα θα αντέξουν. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ναχτεγάλ τώρα. Η κυρία Ναχτεγάλ δεν είναι εδώ όμως. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρολτ. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή που βρήκε μια ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση. Η συμφωνία για τους κανόνες σε ό,τι αφορά τα καλυμμένα ομόλογα εντάσσονται σε μια λογική που θέλει να ενισχύσει την Ένωση Κεφαλαγορών. Είναι ουσιαστικό να μην χάσουμε το στόχο έσχατος σκοπός του νόμου που υθετούμε Στη συγκεκριμένη περίπτωση ουσιαστικά πρόκειται για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας. Βεβαίως προσπαθούμε να φέρουμε στις τράπεζες μια πηγή χρηματοδότησης ε, μακροπρόθεσμη για να ελοπιθεί ο στόχος αυτός. Τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην αποδυναμώσουμε το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών. Καταρχήν, χωρίς αυτό να ε, σημαίνει ότι θα υπάρχει βελτίωση της χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις ε, και τους πολίτες. Και δεύτερον, αν αυτό ενέχει κινδύνους που ε, ουσιαστικά διακυβεύουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι αξιοσημείωτο. Γιατί θα επιτρέψει στις χώρες όπου δεν υπάρχουν ακόμη αγορές αυτές να ευνοήσουν τη δημιουργία ενός ε, εργαλείου ε, που ε, φαίνεται να είναι σταθερό ακόμη και σε περιόδους κρίσης και να φέρθηκε ο συγητής. Άλλα εργαλεία όπως παραδείγματος χάρη μιας ευρωπαϊκής εγγύησης θα συζητηθούν περαιτέρω. Και καθώς τελευταία φορά παίρνω το λόγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω να σας ευχηθώ. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια η κυρία Μπέρες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το πλαίσιο της ελάχιστης εναρμόνισης των εθνικών καθεστώτων που θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι πρόσδεκτο. Θα μπορέσουμε να έχουμε ένα χρήσιμο εργαλείο επαναχρηματοδότησης και θα συνεισφέρει στην εμβάθυση των κεφαλαίων θα πρέπει να θυμηθούμε όμως ε, ότι ε, τα ομόλογα αυτά έχουν επιτρέψει στις τράπεζες να λειτουργήσουν σε δύσκολες συνδικές στην αγορά. Το 2008, την χάρη, όταν είχαμε ε, το, το πόγιο της κρίσης, αυτά παίρνουν τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε εθνική αγοράς. Στη Γαλλία υπάρχει δυνατότητα να ε, έχουμε διαφορετικά στοιχεία κάλυψης. Ε, ε χάρη να έχουμε ε, και ε, δάνεια σε κίνητα αλλά και σε άλλες χώρες Δανία, Σουηδία, Ισπανία ε, και γι' αυτό έχουν εμπνευστεί από τις καλύτερες ε, πρακτικές με την δυνατότητα να έχουμε και αυτή την ευρωπαϊκή ετικέτα. Επίσης επιτρέπει στους πρωταγωνιστές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ετικέτα διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο και μπορούν να ευνοηθούν και οι επενδυτές ακόμη και σε περιόδους ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι τράπεζες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανένα το λόγο για το ΚΑΤΣΔΙ. έτσι λοιπόν θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, για τις ε, παρεμβάσεις σας, ε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία για αυτά τα καλυμμένα ομόλογα. Οι επενδυτές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν ότι αυτά τα χρηματοψηφιακά εργαλεία που αποκαλούνται ευρωπαϊκά καλυμμένα ομόλογα ή premium καλυμμένα ομόλογα, αυτά πάγονται σε ειδική εποπτεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρχει μια ισόρροπη προσέγγιση, να είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν οι βασικές διατάξεις. Ε, βεβαίως, εμείς θέλουμε να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε τα καλυμμένα ομόλογα να γίνουν ακόμα πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρο. Ε, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, για άλλη μια φορά στον ε, συνάδελφο κύριο Λούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συντάλφοι, Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδης ηγητές, κυρίως και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα ήδη ελέγχθησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δύο μόνο παρατηρήσεις θα κάνω. Το πρώτο είναι ένα σύντομο σχόλιο ε, απευθυνόμενες προς τον κύριο Μαριά στον συνάδελφό μου. Βεβαίω και πρέπει κανείς πάντα να εξασφαλίζει ότι τα ομόλογα θα πληρώνονται πίσω. Παράδειγμα, τα κρατικά ελληνικά ομόλογα, παράδειγμα που μερικά δεν αποπληρώνονται. Εδώ όμως μιλάμε για άλλο πράγμα, μιλάμε για ομόλογα τραπεζών. Άρα δηλαδή ε, υπάρχουν εξασφαλίσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πουλ κάλυψης ε, το οποίο είναι προστατευμένο από παρεμβάσεις άλλων ομολογιούχων. Εγώ θα πρότεινα η ελληνική κυβέρνηση στο μέλλον να καταφύγει σε αυτή τη διαδικασία και τα κρατικά της ομόλογα να τα εξασφαλίζει μέσα από πραγματικές αξίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα έτσι ώστε να βελτιωθεί και η αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την δυνατότητα δανειοληψίας. Μετά, Αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, σχετικά ότι δεν είναι καλό να διαταράσει κανείς τις εύρυθμα λειτουργούσες αγορές. Ε, ε, σωστό αυτό, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, γιατί αν δεν θέλει κανείς να διαταράξει καμία αγορά, τότε θα πρέπει να επιτρέπει όλες τις πρακτικές και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει και τις χειρότερες πρακτικές. Αυτό όμως δεν είναι ο στόχος της εναρμόνισης που επιδιώξαμε. Νομίζω τα καταφέραμε καλά να αποφύγουμε αυτόν, τον παραπλανητικό δρόμο. Με πώς με το να προβάλλουμε την ποιότητα της νομοθεσίας σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και με τον τρόπο αυτό ασκούμε πίεση σε άλλα να θελήσουν να προσαρμοστούν. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται γενικά η νομοθεσία για τα καλυμμένα ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό ανοίγουμε ένα πολύ καλό δρόμο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πέντε λεπτά παρακαλώ στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να αρχίσω λέγοντας ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για προφορική ερώτηση τώρα στο τέλος της θητείας, αλλά για ένα παράπονο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώ προ την Επιτροπή και το Συμβούλιο, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει θεμητή συνεργασία, ότι δεν υπάρχει θεσμική συνεργασία ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σοβαρό. Πρώτα απ' όλα θέλω να επενθυμίσω τα γεγονότα. Ήδη το άρθρο 226 της συνθήκης της Λισαβόνας επέτρεψε ήδη από το 2009 όταν εγκρίθηκε η συνθήκη αυτή επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νομοθετική πρωτοβουλία για να ρυθμίζει τις εξουσίες των ερευνητικών επιτροπών. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου σε δύο θέματα, στον εκλογικό ευρωπαϊκό νόμο και στην ρύθμιση ακριβώς των ε, επιτροπών εξέτασης πραγμάτων. Το 2012, τρία χρόνια μετά, από τον David Μάρτεν που ήταν τότε εισηγητή, αρχίσαν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ήδη από την προηγούμενη θητεία δεν υπήρξε συμφωνία και το 2014 σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε το κείμενο αυτό. Εντάξει, χωρί συμφωνία τη Επιτροπή και του Συμβουλίου. Όταν εγώ ορίστηκα εισηγητή στην αρχή αυτή τη θητεία, το 2015, άρχισα να προσπαθώ να κάνω διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για πάνω σε ένα κείμενο το οποίο είχε εγκριθεί από τα θεσμικά όργανα. Και εδώ είναι που αρχίζει το πολιτικό μου παράπονο, γιατί δεν καταφέραμε να πετύχουμε το Σεβούλιο και η Επιτροπή να συνεδριάσουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα θεσμικό τριμερή διάλογο, σε έναν λογικό πολιτικό διάλογο, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο να μα επιτρέπει έναν κανονισμό που να ρυθμίζει τι αρμοδιότητε του σώματο σε θέματα εξέταση των πραγμάτων. Πολλές ε, προσπάθειε κάναμε εμεί με ευελιξία που επιδείξαμε προ την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είπαμε, ετοιμάς, μας είπατε μάλλον ότι είμαστε νέο κείμενο και το κάναμε μετά από εννέα μήνες συνεδριάσεων με τις νομικές υπηρεσίες της Επιτροπής του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τελικά καταλήξαμε σε ένα νέο κείμενο που το ονομάσαμε non-paper. Το παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο και μας απάντησε με επιστολή, όπως κάνει συνήθως, με ενστάσει, νομικέ. Ε, αντιρρήσεις, ανησυχίες. Επί της ουσίας η απάντηση ήταν πάντα επί της διαδικασίας. Κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Μια αποδοχή της διαπραγμάτευσης. Και εξού το παραπονό μας ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν συνεργάστηκαν μαζί μας, δεν θέλησαν να έχουν διάλογο μαζί μας. Και μας ε, ταπεινώσατε κυρίες και κύριοι. Έτσι αισθάνομαι, ειλικρινά και μεγάλη απογοήτευση έχοντας δουλέψει τέσσερα χρόνια με την Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων, με την κυρία Χούμπνερ, για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση που δεν κατέστη εφικτή. Δεν είναι μόνο διαδικαστικό το ζήτημα, κυρίε και κύριοι. Γι' αυτό και έρχεται εδώ το πολιτικό μας παράπονο. Γιατί το πρόβλημα ουσίας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν δέχονται να υπάρχουν επιτροπές με δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων. Όλες αυτές οι εξεταστικές επιτροπές ενοχλούν τους επιτρόπους, ε, τις κυβερνήσεις κλπ. και κλπ. Επί της ουσίας λοιπόν αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι φοβόσαστε. Μήπως κληθούν μάρτυρες, επίτροποι, ε, μέλη κυβερνήσεων. Και αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημα. Δεν θέλετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει μια εξουσία που είναι τόσο σοβαρή όσο είναι οι εξεταστικέ επιτροπές, που είναι κάτι απαραίτητο στον κοινοβουλευτισμό του 21ου αιώνα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να αρνείστε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια δυνατότητα που του έδωσε η συνθήκη τη Λισαβόνα και στον 21ο αιώνα που υπάρχουν τόσα θέματα κακοδίκησης ή που πλήττουν το κράτος δικαίου να μην μπορεί να τα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπούμε απευθείας τους πολίτες για να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν αύριο θα εγκρίνουμε κυρίες και κύριοι ένα ψήφισμα που είναι σκληρό αλλά και δίκαιο. Είναι ένα ψήφισμα ιδιαίτερα επικριτικό απέναντι στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά είναι κάτι αναγκαίο κυρίες και κύριοι. Αυτά θέλω να σας πω. Θα μεταφέρουμε στον ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου και θα του ζητήσουμε στη συνεδριά του με το Συμβούλιο, να το πει θα το στείλουμε στους πίτσεν καντιντάτες από τις διάφορες πολιτικές οικογένειες, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το πολιτικό παράπονο. Και να συζητηθεί αυτό το θέμα και με τους επόμενους. Είναι αναγκαίο προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ένα κοινοβούλιο που να εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματο της Επιτροπής Συνταγματικών Επιθέσεων, η κυρία Χουμπνερ, το ε, κύριο όπλο είναι αυτό για ένα σύγχρονο κοινοβούλιο. Αν σκεφτούμε το Dieselgate, το Panama Papers και άλλα σκάνδαλα, κατανοούμε ότι είναι θεμελιώδες το Κοινοβούλιο να έχει δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων εύρωστο. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη συστηματικά αρνούνται να κάτσουν στο τραπέζι και να κάνουν πραγματική συζήτηση για το περιεχόμενο τη πρόταση του Κοινοβουλίου. Το επιχείρημα ήταν ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου δεν λάμβανε υπόψη τι θεμελιώδει ανησυχίε. Όμω αυτό σημαίνει ότι αγνοείται την ε, ειδική νομοθετική διαδικασία που έχει θεσπιστεί με το άρθρο 226 της ε, συνθήκης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση συμβιβασμού αποδεκτή από όλους. Το Συμβούλιο ζήτησε το αρχική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει ήδη να συμπεριλαμβάνει ένα κείμενο αποδεκτό από το Συμβούλιο. Όμως δεν λειτουργεί έτσι η διαδικασία. Πώς το Συμβούλιο η Κομισιόν θα αντιδρούσαν αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνείται ακόμη και να συζητήσει πιθανούς τρόπους επιτεύξης συμφωνίας παραδείγματο χάρη στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντα την πρόφαση ότι δεν του αρέσει η πρόταση τη Κομισιόν. Επιπρόσθετα, η στάση αυτή δεν είναι συμβατή με την αρχή τη ειλικρινού συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων που όλοι πρέπει να σεβόμαστε. Εδώ διακυβεύεται ένα θεμελιώδες θέμα σεβασμού για τα προνόμια του Κοινοβουλίου και για την θεσμική ισορροπία. Πρέπει το Συμβούλιο και η Κομισιόν να το κατανοήσουν και τελικά δεν έχουμε υποχρέωση να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, αλλά έχουμε το καθήκον να προσπαθήσουμε. Δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν ανταπεξέλθει στο καθήκον αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Τσιάμπα εξ ονόματο του Συμβουλίου. Αγαπητέ Πρόεδρε, πλησιάζει το τέλος της θητείας και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε το σημαντικό θέμα της άσκησης ε, του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων του Ευρωκοινοβουλίου. Καταρχάς να σας πω ότι συμφωνούμε ως ε, Συμβούλιο ότι οι εξεταστικές επιτροπές είναι ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί το πολιτικό έλεγχο στην Ένωση και αυτό κατοχυρώνεται στο σεβασμό της ε, αρχής της δημοκρατίας ε, του κράτους δικαίου όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Μετά την έκθεση του 2011 εξετάσαμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου διάφορες προτάσεις με πολύ επικοδομητικό πνεύμα και πάντοτε με την ειλικρινή συνεργασία ως βάση. Είναι γνωστό όμως ότι σε αυτή την έκθεση, την έκθεση Μαρτή υπάρχουν σοβαρές θεσμικές επιφυλάξεις ε, και από πλάσκο και Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το 226 το άρθρο αυτό της συνθήκης ε, και σε ό,τι αφορά την επέκταση των εξουσιών και δικαιωμάτων ε, των, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεωρείται ότι αντιβαίνει στο άρθρο 226 παρά τις προτάσεις συμφιλίωσης διαφόρων επιλογών ζητημάτων Παραδείγματο χάρη, οι εμπειρογνώμονε των νομικών υπηρεσιών προσπάθησαν και με πολλέ συναντήσει έχουμε κάνει πρόοδο σε κάποιε μη προβληματικέ διατάξεις, αλλά δεν έχουμε λύσει τα πιο πολύπλοκα ζητήματα νομικού και πολιτικού χαρακτήρα όπως αναφέρεται σε επιστολή που απεστάλλει στην ε, κυρία Χούπνερ πέρυσι τον Οκτώβριο 25 του μήνα συγκεκριμένα από την Προεδρία του Συμβουλίου. Καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεσης ε, κυρίου Χαουρέγγι Ορτουόντο ε, για την αναζωγόνηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Είναι ένα non-paper αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμένε βελτιώσει σε σχέση με τι προτάσει του 2014 και ορισμένε από τι ανησυχίε του Συμβουλίου διασκεδάζονται και γίνονται κάποιες προτάσεις ε, όπως πρότειναν νομική υπερονόμηση των τριών θεσμικών οργάνων. Όμως αυτό ήταν επίσημα έγγραφο. Ξεκολουθεί να περιλαμβάνει κάποιες διατάξεις που θα γύρουν σημαντικά πολιτικά και θεσμικά ζητήματα. Το έχουμε πει και ξαναπεί και κατά το παρελθόν. Επί της ουσίας η θέση μας για τα θεμελιώδη ζητήματα δεν έχει αλλάξει μετά την 6 η Μάρτη και για να είμαι πιο συγκεκριμένος θα ήθελα μεταξύ των πλέον προβληματικών ζητημάτων να αναφέρω ότι γίνεται με κάποιους που καλούνται ως μάρτες και δεν είναι ε, υπάλληλοι, ε, οι αξιωματούχοι. Κροάσεις τέτοιων μαρτύρων η εξουσία να ζητηθούν έγγραφα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ρόλο στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Και τέλος, η διατάξη για τις κυρώσεις είναι κάποια θέματα που μας απασχολούν στο ποινικό δίκαιο. Είναι θέματα που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως και ε, στο πλαίσιο του κώδικα ποινική δικονομίας. Δεν θα έλθω, επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι γνωρίζετε πολύ καλά τις ανησυχίες του Συμβουλίου, όπως αναφέρονται άλλωστε λεπτομέρειες και στην επιστολή που προανέφερα. Από την αρχή της Προεδρίας μας προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις ε, ε, και σε επίπεδο κομισιών. Είχαμε πολλές άτυπες επαφές και οι ε, προκάτοχοι μου ε, συνάντησαν τον κύριο Χαουρέγγι και την κυρία Χούμπνερ και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε να είμαστε ανοιχτοί ε, προ οικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να, να στήσουμε ε, μια διέξοδο ε, σε σχέση με το πολύπλοκο αυτό ζήτημα. Αν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει το έργο με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, είμαστε και εμεί έτοιμοι να το κάνουμε με πλήρη σεβασμό στην αρχή τη ειλικρινού συνεργασία. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Να παρακαλέσω την Επίτροπο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι βουλευτές, ε, Χαίρομαι που με την προφορική ερώτηση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα ε, από πλευρά τη Κομισιόν να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά το Κοινοβούλιο διατυπώνει πρόταση, αλλά με τη διαδικασία απαιτείται συγκατάθεση Συμβουλίου και Κομισιών. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε συγκεκριμένε προτάσει για μια τέτοια ρύθμιση, ένα τέτοιο κανονισμό και ανεπίσημα είχαμε αυτό το non-paper τελευταία, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πέρυσι τον Απρίλιο και διαβιβάστηκε σε Συμβούλιο και Κομισιόν πέρυσι τον Μάιο. Αναγνωρίζουμε πως η μια ανεπίσημη πρόταση ε, έχει καταρτιστεί ε, με πιο συγκεκριμένου όρου και περιλαμβάνει αρκετές βελτιώσεις. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες για τη συγκρότηση μιας εξεταστικής επιτροπής, οι διαδικαστικοί κανόνες που έχουν να κάνουν με την έρευνα ή τη δημιουργία ενό κεντρικού ε, συνδέσμου. Είναι θετικές εξελίξεις. Ναι, επίσημη πρόταση επίση περιλαμβάνει αναφορά ε, σε έναν κανονισμό για την ε, προστασία φυσικών προσώπων σε ό,τι την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και λαμβάνει υπόψη και τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Ωστόσο, αυτό το ανεπίσημο έγγραφο εξακολουθεί να δημιουργεί κάποιε νομικέ και θεσμικέ ανησυχίε που ήταν και στο επίκεντρο των συζητήσεων ε, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου από το 2012 και οι πιο βασικέ από αυτέ τι ανησυχίε είναι οι κυρώσει για τη μη συμμόρφωση με τι διατάξει του κανονισμού ορισμένε πτυχέ ε, των εξαστικών μέσων και εργαλείων που θα έχουν στη θέση του αυτέ οι επιτροπέ, επιτόπιε, έρευνε, ακρόαση με επιτρόπους νυν και τέο, με ακρόαση με υπαλλήλου νυν και τέο και τα φυσικά πρόσωπα που είπαμε. Επίσης, ε, μισάγεται ένα νέος κανόνα για τα 11 μέσα, περίπτωση παραβίαση των διατάξεων της συνθήκης από μια εξεταστική επιτροπή, από τα μέλη τη, από παλίλου, εξωματούχου ή άλλε υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τέλο, υπάρχουν κάποιε διατάξει που από ό,τι φαίνεται δίνουν διακριτική ευχέρεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την αναστολή των διαδικασιών τη εξεταστική επιτροπή ε, όταν είναι στο δικαστήριο η διαδικασία. Παρά ε, και με επιφύλαξη αυτέ τι ανησυχίε, θέλω να πω ότι εμεί ε, είμαστε διατεθειμένοι ω Κομισιόν να συνεχίσουμε οικοδομητικέ τριμερίε συζητήσεις ε, με στόχο την εξέβρεση των κατάλληλων λύσεων ε, σε ό,τι αφορά τι αποκλήσει που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Μελλοντικό ε, κανονισμό σε ό,τι αφορά το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκέ εργαλείο που θα σέβεται και τα θεσμικά προνόμια αλλά και των νομικά πλαίσια των κρατών μελών. Αυτό είναι ο στόχο μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε, ο κύριος Βίλαν δεν είναι στην αίθουσα που θα έπρεπε να λάβει το λόγο. Ως εκ τούτου, εκ μέρους των ε, φιλελευθέρων, η κυρία Γουαρακουτού. Α, η κυρία Ρουΐς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν μας ακούσατε, κυρία Τσάμπα. Σας είπαμε. Πολλάκι. Καθ' όλα αυτά τα έτη και το είπε και ο κύριος Χαουραγκή, ότι μιλάμε για έλλειψη συνεργασίας. Δεν υπήρξε πιστή συνεργασία. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό το κοινοβούλιο μας έλειπαν ε, ικανότητες κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας για να μπορέσουμε να εργαστούμε καλύτερα στην περίπτωση των Panama Papers και στο Diesel και στην Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία γιατί εσείς θελήσατε να μπλοκάρετε αυτή τη δυνατότητα. Αν ο κύριος Χαουρέγγι έχει στο DNA του τη διαπραγματευτική ικανότητα και <laughs> μπορεί πολύ εύκολα να φτάνει συμφωνίες και δεν μπορούσε να το κάνει, είναι επειδή δεν υπήρξε συνεργασία από εσά. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους λοιπόν. Εδώ και 25 χρόνια λειτουργούμε με μια απόφαση η οποία είναι μικρή και παροχημένη. Αυτό δεν είναι το Κοινοβούλιο του 1995. Χρειαζόμαστε αυτά τα προνόμια τα οποία εσείς ε, φέροντας διάφορα επιχειρήματα και διάφορους λόγους δεν θέλετε να δώσετε σε αυτό το κοινοβούλιο και κάνετε λάθος γιατί χάνουμε αξιοπιστία, γιατί πρέπει να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα εξέτασης πραγμάτων δεν είναι δίκαιο, δεν είναι αξιοπρεπές αδελφά θεσμικά όργανα, όπως είναι το Συμβούλιο και η Κομισιόν, να δένουν τα χέρια του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Όταν ε, ασκούμε τα καθήκοντα που μας ε, έχουν δοθεί. Εμείς αυτό το καθήκον έχουμε να υλοποιήσουμε. Δεν είναι δίκαιο ο κύριος Χαουρέγγι να έχει εργαστεί για πέντε χρόνια όπως το έκανε και η πρόεδρος της ε, Κομισιόν της Επιτροπής Συγγνώμης Συνταγματικών Επιθέσεων, η κυρία Ντέντα Χνούμπλερ και η γραμματεία της ΑΦΚΟ. Δεν είναι δίκαιο Μα κλείσατε την πόρτα στα μούτρα. Έτσι λοιπόν το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν ε, υπήρξε ε, ιδέους επιμέλεια από την πλευρά σας και ευχαριστώ τον κύριο Χαουρέγγι και πάλι ε, για όλο του το έργο του. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα δεν βλέπω τον κύριο Σόλτς, ο οποίος θα έπρεπε να πάρει το λόγο εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Έτσι λοιπόν, να ακούσουμε την κυρία James, εξ του EFDD. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε χρειαζόταν απόδειξη ότι ε, τελικά ε, αποτελεί ένα προπέτυσμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημοκρατία. Το έχουμε εδώ. Αν πρέπει να έχει νόημα η δημοκρατία, τότε οι νόμιμοι επλαγμένοι, οι βουλευτέ εδώ, θα πρέπει να επιτρέπεται να αμφισβητούν οτιδήποτε. Ε, αφορά αυτούς που εκπροσωπούν. Το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων ε, θα έπρεπε να έχει νομική υπόσταση. Διαφορετικά ποιο είναι το νόημα. Δείχνεται ότι απλώς μια μαριονέτα είναι το Κοινοβούλιο ε, για όσους στην Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν έχουν εκλεγεί. Αυτή ε, η νομική υπόσταση, αν δεν αναγνωριστεί, αυτό υπονοείται και με ενοχλεί που το Συμβουλίο και η Κομισιόν λειτουργούν με έναν τρόπο παρακόλλησης όταν μιλάμε για τη διαφάνεια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, αναρωτιέται η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι λαϊκιστέ και οι ευρωσκεπτικιστέ ανθίζουν και ευημερούν. Έχετε την απάντηση ενώπιον σα. Μιλάμε για ε, ένα μεγάλο πλήγμα στη δημοκρατική διαδικασία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Ποσπισίλ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λυπούμε πολύ με τη θέση του Συμβουλίου και της Κομισιόν, διότι με το πρωτογενές δίκαιο έχουμε σαφές, ξεκάθαρο δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων. Και αν αυτό ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί μέσω εκτελεστικού κανονισμού, πραγματικά είναι ντροπή. Με εντυπωσιάζουν δε περισσότερο, θα έλεγα, ε, τα όσα είπε το Συμβούλιο, η συμπεριφορά του Συμβουλίου. Δεν μπορώ να την κατανοήσω. Θα περίμενα από εκπρόσωπο ενός δημοκρατικού κράτους μέλους να κάνει περισσότερα για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε οι άμεση εκλεγμένοι πρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε εξουσίες, τις οποίες μας εκχωρεί το βασικό δίκαιο, το πρωτογενές δίκαιο και δυστυχώς Συμβούλιο και Κομισιόν μειώνουν τις δυνατότητες που έχουμε και την εξουσία μας. Αν αυτό συνέβαινε κάπου αλλού θα το καταλάβαινα, γιατί πολλές φορές ε, ασκούμε κριτική σε τρίτες χώρες και στον τρόπο με τον οποίο παραβιάζεται το δίκαιο όμως εδώ έχουμε ήδη στη δική μας την πίσω αυλή το ίδιο πρόβλημα. Παρακαλώ λοιπόν σκεφτείτε το, προσπαθήστε τουλάχιστον, διότι πρόκειται για ε, κάτι που πραγματικά μας δυσφημεί. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ στη διαδικασία προσέλκυσης ε, της αποσύγησης του Μαριάς ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός κοινοβουλίου η νομοθετική λειτουργία ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και οι εξεταστικές επιτροπές. αυτά κάνουν τα δημοκρατικά κοινοβούλια και το δικαίωμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου να προχωρεί στην εξέταση πραγμάτων δηλαδή να κάνει εξεταστική επιτροπή προβλέπεται αυτοτελώς από το πρωτογενές δίκαιο επομένως πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξασκεί αυτά τα καθήκοντά του διότι όταν δεν προχωρά σε εξεταστικές επιτροπές όταν έχουμε σκάνδαλα όπως τα luxleaks τα panama papers το diesel σκάνδαλο και δεν κάνει τίποτε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τότε μειώνεται η αξιοπιστία του δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις του με τους πολίτες αυτό το δικαίωμα θέλουμε να εξασκούμε αυτοτελώς αυτό διεκδικούμε και νομίζω ότι η τοποθέτηση του συμβουλίου δεν συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Ήρθε ο κύριος άρα μπορώ να του δώσω το λόγο για 1,5 λεπτό εκ μέρους τη ομάδας της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα χθε εξ αρχή να σα πω ότι εγώ είμαι υπέρ ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πλέον, διότι από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μα δικαστικώ. Κατά την άποψή μου, είμαστε και υποχρεωμένοι ω προ αυτό, διότι είμαστε το Κοινοβούλιο των Ευρωπαίων Πολιτών, των Ποτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το δικαίωμα ε, αυτό είναι δικό του. Να έχουν δηλαδή ένα ισχυρό κοινοβούλιο που οι προνομίε του να γίνονται ε, σεβαστέ. Ε, υπάρχει παρελκυστική πολιτική από το Συμβούλιο και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι που ασκούν επιρροή στα μεγάλα πολιτικά κόμματα και οι οποίοι φοβούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δηλαδή καλεί κάποιους, ε, κάποιο μέλη κυβερνήσεων των κρατών μελών ή συγκεκριμένους ε, μάρτυρες, τι πρόβλημα υπάρχει. δεν θα πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες αυτών των εξεταστικών επιτροπών και τι γίνεται εάν δεν γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ο θεματοφύλακα τελικά των συνθήκων. Είναι στην ίδια πλευρά με το Συμβούλιο. Ε, και ε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ε, πώς το ακούν αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή ε, οι επιτροπές, παραδείγματο χάρη εξεταστικές του Κοινοβουλίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους ε, τα έγγραφα τα οποία ζητούν. Τι έχετε να κρύψετε, τι θα σκεφτεί ο κόσμος όταν ακούσει. Ε, δεν είναι ε, περίεργο να μην έχετε την ε, ευθύνη να δώσετε κατάθεση. ευχαριστώ πολύ. Ναι. Το λόγο έχει τώρα η Επίτροπος κυρία Μπιενκόφσκα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τα αξιότιμα μέλη για τις παρατηρήσεις που έκαναν. Θα ήθελα να επαναλάβω το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο που δραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο. Απότερο στόχο είναι τα συμφέροντα και ανησυχίε των πολιτών όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου να αντιμετωπίζονται σωστά, να διασφαλίζεται αυτό. Αναγνωρίζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο που έχουν κάνει τα θεσμικά όργανα και αναγνωρίζει ότι το ανεπίσημο έγγραφο αντιστοιχεί σε σαφή πρόοδο σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις. Από την άλλη όμω, όπως είπα και νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ανεπίσημη αυτή πρόταση έχει ακόμα κάποια θεσμικά και νομικά κενά, όπως για παράδειγμα οι κυρώσει τα ένδικα μέσα τα οποία προβλέπονται και το καθεξής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο εργαλείο το οποίο να τηρεί τα βασικά θεσμικά προνόμια των κρατών μελών αλλά και των θεσμικών οργάνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν ε, οι κατάλληλε τριμερεί διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασκεδαστούν οι ανησυχίε, οι οποίοι ακόμα υφίστανται. Ελπίζω ότι στο πολιτικά αυτό αλλά σημαντικό θέμα θα σημειωθεί, ελπίζω θα σημειωθεί πρόοδος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Τσάμπα, ο υπουργό. Παρακαλώ conclude, Κατακλείδη. Να ευχαριστήσω όλους για την ανταλλαγή απόψεων. Ξεκαθαρίσαμε τις θέσεις μας, εκατέρωθεν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι προηγούμενες προεδρίες έδειξαν ανοιχτό πνεύμα εν ώψη της προσπάθειας εξέβρεσης λύσης. Συζήτησαμε το θέμα σε βάθος στην αρμόδια ομάδα εργασία. Δυστυχώ, υπό τι παρούσες συνθήκε, είναι σαφέ ότι δεν είναι δυνατόν να κλείσει ο φάκελο στη διάρκεια της παρούση θητεία του Κοινοβουλίου. Για άλλη μια φορά όμω, το Συμβούλιο σα διαβεβαιώ είναι ταγμένο στην προσπάθεια συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά τον Μάιο. Είναι προ το συμφέρον όλων, να θεσπίσουμε ενημερωμένους κανόνες, να επερμηθούμε του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εξαίρεση των πραγμάτων. Ευχαριστώ λοιπόν τον κ. Ντόντοφ για τη σπουδαία δουλειά που έκανε ο συγητής. Ξέρω ότι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βελτιώσει την τελευταία έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για άλλη μια φορά. Είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται η Προεδρία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία που είχαμε τους τρεις τελευταίους μήνες. Είχαμε ειλικρινή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για εμάς ήταν ε, χαρά να συνεργαστούμε με την Ρουμανική Προεδρία, λέει ο Πρόεδρος. πρόεδρος συνεχίζει. Έλαβα σχέδιο ψηφίσματος στο τέλος της συζήτησης. Το υποβάλλει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια αύριο. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a to jest sprawozdanie pana Fernandesa i pana Guiteliego. Επόμενο σημείο, Φερνάντε Γκολτιέρη, έκθεση σχετικά με την πρώτη κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη θέσπιση του προγράμματο InvestEU. Δίνω τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Φερνάντε. Κύριε Πρόεδρε, χαιρετώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ όλες και όλους που εργάστηκαν επί του θέματος που αφορά την περίοδο 2021-2027. Ευχαριστώ και τον ε, Ρομπέρτο Γαλτιέρη, ο οποίο ε, και αυτό εργάστηκε σκληρά. Και να ευχαριστήσω επίση θερμά τους συναδέλφου που εργάστηκαν σκληρά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το σχέδιο Juncker, το ταμείο Juncker. Ευχαριστώ τους και και τους εργάτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και την Γραμματεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Την περιοδο 2020 έχουμε μπροστά μας έναν μηχανισμό ο οποίος ε, συγκεράζει και απλουστεύει τη λειτουργία 14 χρηματοδοτικών μηχανισμών. Ενοποιούνται και απλουστεύονται. Χρειάζεται όμως ε, για να γίνει κάτι τέτοιο ένα φιλόδοξο όραμα. Όπως είπα Έχουμε σύμπηξη 14 διαφορετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών και όλα αυτά με τη μορφή εγγύσεων 40,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιήσουν συνολικά περίπου 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια μικρή διαφορά μεταξύ 650 που θέλει το Συμβούλιο. Ε, εν πάση περιπτώσει έχουμε συμφωνήσει όλα με την εξαίρεση αυτού Χαίρομαι, εν πάση περιπτώσει, για αυτήν την προσωρινή συμφωνία. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σύντομα. Πρόκειται λοιπόν για το νέο ταμείο Invest εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε τέσσερις θηρίδες, κατά κάποιο τρόπο, επενδύσεις σε αϊφοροανάπτυξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τρίτον έρευνα και καινοτομία και τέταρτον, τέταρτος άξονας, κοινωνική στόχη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εξομαλύνει τις διαφορές σε επενδύσεις μεταξύ περιφερειών. Πρέπει οι διακρίσεις, οι διαφορές να εξελιχθούν και όλοι να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα τα κρατημέλη πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν ένα νέο πεδίο διότι τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και αυτά στις χρηματοδοτήσεις εθελοντικά μπορούν να βοηθήσουν για παράδειγμα επενδυτικές τράπεζες σε κάποιο άλλο κράτος μέλος στην περίπτωση που παρατηρούνται αδυναμίες. Η κάθε χώρα λοιπόν πρέπει να κάνει αυτό που της αναλογεί. Πρέπει επίση οι διάφοροι οργανισμοί χρηματοδότηση αναπτυξιακή μορφή να προετοιμαστούν. Εμεί βλέπουμε το θέμα θετικά. Θέλουμε να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε θέσει εργασία ποιοτικέ. Θέλουμε καλύτερη διακυβέρνηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών. Και πέραν αυτού όσον αφορά το συμβουλευτικό